Το πρώτο θέμα αφορά την έκθεση της κυρίας Ρέγνερ και την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Στίβ Μπριουά. Ο κύριος Κόμπεν ζήτησε το λόγο για διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζω και ανησυχώ τα μάλα, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε ασυλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε φορά όμως ε, συζητούμε αιτήσει για άρση της ασυλίας ευρωβουλευτών. Δεν με ενδιαφέρει αν ε, είναι φασίστας, κομμουνιστής, δημοκράτης ο ενδιαφερόμενος. Αλλά θα προασπίσω τα δικαιώματά τους. Και αν συνεχίζουμε να έρουμε ασυλίες, θα εκενώσουμε περιεχομένου την ε, έννοια της ασυλίας. Και δεν έχει νόημα να μιλάμε ελεύθερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν προστατευόμαστε με την ασυλία για αυτά που λέμε. Δεν θα πρέπει συνεχώς να έρουμε την ασυλία ευρωβουλευτών μόνο επειδή είναι κάποιο μέρος του Εθνικού Γαλλικού Μετόπου, του Front National, δεν είναι αρκετός λόγος για να έρουμε την ασυλία του. Σας διαβεβαιώ κύριε Κόμπερν ότι η συζήτηση και η σχετική ακρόαση έγινε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια. Σημειώνω αυτά που είπατε, αλλά θα ψηφίσουμε Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Τσόκα για τη Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας. Θα γίνει με ονομαστική κλίση. Ψηφοφορία είναι θέμα συνένεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η σύσταση Τζόκα. Επόμενο θέμα αφορά τη σύσταση ειδική Επιτροπής ε, για τα φυτοφάρμακα και τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, τις αρμοδιότητες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της. Ψηφίζουμε Διανατάσσω τη χειρός. Ποιος είναι υπέρ τη σύσταση αυτής τη ειδική επιτροπή Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Φοντίνων Χόχενστάιν για το γεωγραφικό αποκλεισμό και τις άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ηθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών. Ψηφίζουμε πρώτα δύο τροπολογίες, τις 67 και 68, πανομοιότυπες για την απόρριψη πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ε, προ... Προσωρινή συμφωνία. Τροπολογία 70 της Επιτροπής. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τροπολογία 69. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Gerling για τι οικονομικά αποδοτικές μειώσει των εκπομπών και παιδείς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Θα ψηφίσουμε πρώτα την προσωρινή συμφωνία, την τροπολογία δηλαδή 166, ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και τις δηλώσεις της Επιτροπής, τροπολογία 167. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνονται. Οπότε ολοκληρώσαμε την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περνάμε στην έκθεση Ζωνάς Φερνάντες ε, με θέμα την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016. Θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε την παράγραφο 2, αρχικό κείμενο, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 13. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Παράγραφος 26. Αρχικό κείμενο. Α, συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Παράγραφος 18. Τροπολογία 9 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της 18 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της παραγράφου 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 18 με ονομαστική κλίση και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση. Με ονομαστική κλίση, τροπολογία 10, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 26. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτω. Αρχική παράγραφος 27 σε τρία τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Διανατάσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχική παράγραφος 31 με ονομαστική κλίση, της ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 32 σε τρία τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τρίτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 35, αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 38, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 40, τροπολογία 17 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 44, ε, τροπολογία 12, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 45. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 46. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα ονομαστικά το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Φερνάντες. Και περνάμε στην έκθεση Μπούζεκ με θέμα την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ε, με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μπούζεκ. Ολοκληρώσαμε το χρόνο ψηφοφορίας. Να σας ζητήσω παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα για να προχωρήσουμε στις αιτιολογίες της ψήφου.